στο ελεγκτικό συνέδριο και στα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των δημοσίων δαπανών σε όλη την Ευρώπη από κοινού. Ευχαριστώ. Μπενόβα. Κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα.